θα μάθατε μάλλον τα λυπηρά γεγονότα τη επιθέσεω του Σαββατοκύριακο στην Βόρειο Ιρλανδία εναντίον μιας Βρετανικής βάσης που ε, κόστη τη ζωή σε δύο στρατιώτε από το Birmingham και το Λονδίνο και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ε, ατόμων μεταξύ των οποίων οι δύο ήταν και πολίτες και μάλιστα ο ένας ε, Πολωνός πολίτης επιθέσεις κατά των δυνάμεων ασφαλείας στη Βόρεια Ιρλανδία είναι μια φρικτή πράξη και την καταδικάζω με τον πλέον απερίφραστο τρόπο. Our sympathies the families. Εκφράζουμε τα αυτά συλληπιτήριά μας προς τις οικογένειες και τους οικείους ε, των ε, των στρατιωτών που θυσίασαν τη ζωή τους για την συμφιλίωση των κοινοτήτων, ε, για την ευημερία των κοινοτήτων αυτών, καθώς και των άλλων ε, θυμάτων. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση στη Βόρεια Ιρλανδία από 12